η συνδιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 134 του κανονισμού να συγκαλέσει έκτακτη ολομέλεια στις 23 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, 3 με 5 το απόγευμα. Στην έκτακτη αυτή ολομέλεια θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Βαν Ρόμποϊ, και θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Κίνς. Uh, Κύριος Άτκινς, συγγνώμη. Διαδικαστικό. Θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Δηλαδή θα βρίσκουμε Στη γραφεία μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αιτήσει ε, που μας ζητούν να ψηφίσουμε και ψηφίσματα που ζητούν την ε, υπογραφή μας. Αυτά είναι σκουπίδια και δεν ελέγχουμε αυτή τη ροή τέτοιων ε, σκουπίδιων στα γραφεία μας. Θα ήθελα πραγματικά να μπει ένα τέρμα. All right, Atkins, we take good note. Καλώς, το σημειώνουμε κύριε Άτκινς. Σημειώνουμε αυτή την παρατήρηση, διαμαρτυρία, ό,τι τέλος πάντων είναι αυτό που είπατε. Yes, Mr. Lange. Ο κύριος Για το ίδιο διαδικαστικό θέμα δεν αρκεί να το σημειώσει ο Πρόεδρος. Εγώ απαιτώ να σταματήσει αυτή η πρακτική. La presidencia η Προεδρία το σημειώνει και θα λάβει τα δέοντα μέτρα. Αλλά πρώτα πρέπει να το σημειώσει και μετά να λάβει τα μέτρα, τα κατάλληλα. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρίσατε στο Κοινοβούλιο μία αντιπροσωπεία της ε, Εθνικής Βουλής του Κουβέιτ στο Προεδρείο των Επισήμων. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την αντιπροσωπεία από το Κουβέιτ, από την Κουβετιανή Βουλή. Está, presidida por el señor...